Παρακαλώ να καθίσετε στις θέσεις σας. Ξανασυνεχίζουμε τη συζήτηση, κυρίε και κύριοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα το πρωί μάθαμε συγκλονιστικές ειδήσει από το Πακιστάν. Σε ένα σχολείο έχασαν τη ζωή τους 120 άτομα και περισσότερα, από τα οποία Εκατό ήταν παιδιά. Τα δολοφόνησαν κατά αποτρόπαιο τρόπο οι Ταλιμπάν. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι βρέθηκαν υπό την... Ε, πολύ περισσότεροι ήταν αυτοί οι οποίοι βρέθηκαν υπό τον έλεγχο των τρομοκρατών αυτών. Μα συγκλονίζει το γεγονός και δείχνει για άλλη μια φορά τον απάνθρωπο τρόπο με τον οποίο οι Ταλιμπάν προσπαθούν με τρόπο αποτρόπαιο, με απάνθρωπο τρόπο να επιβάλλουν την ιδεολογία τους. Και αυτό που πάνω απ' όλα μας συγκλονίζει είναι ότι δεν δίστασαν να δολοφονήσουν και παιδιά. Οι σκέψεις μας είναι στις οικογένειες, τους φίλους των παιδιών αυτών. Είμαστε στο πλευρό του Πακεριστανικού λαού και εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκφράζω τα βαθύτατα συλληπιτήριά μας σε όλους τους συγγενεί και υγιούς των θυμάτων. Και εύχομαι